Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Ο εκπρόσωπος της Προεδρίας, ο κύριος Πέτερ Νέτσας, ο Επίτροπος Όλη Ρεν, βρίσκονται εδώ. Αγαπητέ εισηγητή, αγαπητοί συνάδελφοι, με μεγάλη χαρά σήμερα το απόγευμα θα ασχοληθούμε με δύο πολύ σημαντικά πακέτα, το πακέτο των κλιματικών αλλαγών και το πακέτο που αφορά την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από τη συνεργασία μας με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγκρίνοντας λοιπόν αυτή την πολιτική καταδεικνύουμε ότι μπορούμε να αναλάβουμε δραστηριότητα σε τομείς κλειδιά όπως την βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές. Έτσι υποστηρίζουμε την σημασία της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας υπέρ των πολιτών ως προς το πακέτο των κλιματικών αλλαγών έχουμε εδραιώσει το πρωτογενές δίκαιο για να φτάσουμε στους στόχους μας μέχρι το 2020 για να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο. Αυτό θα μας βοηθήσει επίσης να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να μειώσουν τις εκπομπές θερμοκηπίου. Ο οι συγητής, μάλλον οι συγητές, Ντόιλ και Χάση που βρίσκονται μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Βλέπω ότι η κυρία Χάση είναι εδώ, η κυρία Ντόιλ ίσως να μην έχει φτάσει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει θα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε και νέες τεχνολογίες και αποθήκευση του άνθρακα, δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Έτσι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην διάσκεψη της Κοπενχάγης το Δεκέμβριο φέτος για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την αξιόπιστη πολιτική μας. Σε σχέση με την ασφάλεια στη θάλασσα, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και το Κοινοβούλιο έφτασαν σε συμφωνίες μετά από σκληρή δουλειά εδώ και τρία χρόνια. Και αυτό αποδεικνύει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι σε θέση να βοηθήσει για την ε, πρόληψη και για να ε, μπορέσουμε να αποφύγουμε ατυχήματα όπως του Έρικα και του Πρεστίζ στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι πάρα πολλές από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαμέσου της ε, προσωρινής επιτροπής Αυτά έγιναν νόμος και μετά από τον έλεγχο και την εποπτεία στα πλοία και τις θαλάσσιες μεταφορές βλέπουμε ότι η ασφάλεια θα βελτιωθεί και επίσης θα τονίσουμε αυτούς τους τομείς σε σχέση με τις έρευνες και την απόδοση ευθυνών. Αυτά όλα θα μας τα πει η κυρία Ντόιλ όταν φτάσει Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος στην Τσεχική Προεδρία το Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και τις Επιτροπές Μεταφορών και Βιομηχανίας, τους Προέδρους τους και όλους όσους συνεισέφεραν σημαντικά σε αυτό το τομέα και θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς που ήσασταν παρόντες όταν υπογράψαμε αυτή, αυτή την πράξη σήμερα το απόγευμα, αυτή την ομοθετική πράξη. Υπάρχουν και δύο επικεφαλής ομάδων που βρίσκονται μαζί μας ε, σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα τώρα ο εκπρόσωπος της Αιχικής Προεδρίας να λάβει το λόγο. Eh, eh. Κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω διότι με καλέσατε σε αυτή την σύνοδο